μέτρο για την εφαρμογή της οδηγίας στην επικράτειά τους και παρακολουθώ εκ του σύνεκης εξελίξεις και στα λοιπά κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Πέρα στη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Έκθεση του κυρίου Χέκμαρκ για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο η συγκεκριτής. Βρισκόμαστε μπροστά σε θέματα και συναντήσει κέρια σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και την παγκόσμια οικονομία. Αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την επόμενη εβδομάδα η λέσχη των 20 στις Κάνες θα αποφασίσουν σημαντικά θέματα. Αυτή η έκθεση θέλει να υποβάλει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη συνάντηση της Λέσχης των 20, G20. Είναι μια συνάντηση που θα διαξαχθεί σε μια συγκυρία πολύ σημαντικών και δύσκολων προβλημάτων παγκόσμια, αλλά και εξίσου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο παγκόσμια. Είναι επίση μια συνεδρίαση, μια συνάντηση που θα αντιμετωπίζει το γεγονό ότι η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίζεται από ανισόρροπες, μη ισόρροπε σχέσεις και θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε πλεονασματικέ χώρε και ελληματικέ χώρε. Πίσω από αυτή την εικόνα αποκρύπτεται το γεγονό ότι έχουμε και μία σειρά αναδυόμενων οικονομιών που έχουν συνεισφέρει σε αλλαγέ στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Και βλέπουμε εδώ και θέματα φτώχεια, αλλά έχουμε ακόμα και αρκετές χώρες ε, που πλήττονται από την φτώχεια και που χρειάζονται μεγαλύτερες ευκαιρίες για, ευκαιρίες για πρόοδο και ανάπτυξη. Βλέπουμε και τις πολιτικές που ακολουθούνται από κάποιες ε, μεγάλες οικονομίες μεγάλων χωρών που συνεισφέρουν στις μη ισορροπές σχέσεις. Ε, απουσία ανταγωνιστικότητας σε άλλες χώρες προσθέτουν και αυτό και προσθέτει και αυτή ως στοιχείο στα προβλήματα. Πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να εξευρεθεί μια ισορροπημένη, ισόρροπη σχέση. Χρειαζόμαστε την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και τα αντίστοιχα σωστά θεσμικά όργανα γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι σε χώρες με έλλειψη ανταγωνιστικότητας και σε περιοχέ και περιφέρειε χωρί ανταγωνιστικότητα χρειαζόμαστε νέε πολιτικέ και μεταρρυθμίσει. Ταυτόχρονα όμω χρειαζόμαστε την διασφάλιση των εμπορικών ροών προς αυτές τις αναδιόμενες ε, οικονομίες ε, που σήμερα προστατεύονται με τεχνητές ε, νομισματικές πολιτικές. Στην έκθεση που έχει τύχει ευρύτατης υποστήριξης στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τους σκιώδεις εισηγητές που κατέστησαν εφικτό να εξευρεθούν ευρέως αποδεκτοί συμβιβασμοί. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις διαρθρωτικές ε, δυσαναλογίες και ασυμμετρίες και να δούμε τα αίτια των μη ισόρροπων σχέσεων. Πρέπει να διασφαλίσουμε σε παγκοσμιοποιημένο επίπεδο εποπτεία που θα είναι αποτελεσματική και πρέπει να επιτύχουμε πολιτικές που, ε, και ε, νομισματικές πολιτικές που θα είναι μετατρέψιμες και θα επιτρέπουν μεγαλύτερες συναλλαγές όσον αφορά τις πλεονασματικές χώρες και τις ελληματικές χώρες. Είναι σημαντικό όμως να δούμε και την θεσμική αρχιτεκτονική και όσο περισσότερο χρειαζόμαστε αυτή την οικονομική, οικονομική διακυβέρνηση <clears throat> θα πρέπει να αυξηθεί η ανάγκη λογοδοσίας, διαφάνειας <clears throat> και της εμπλοκής και αρχιτεκτονικής δομής θεσμικών οργάνων. Πιστεύουμε ότι η λέσχη των 20 οπωσδήποτε είναι μία από τις πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές, μία από τις πιο σημαντικές δομές. Πρέπει όμως και είναι εξίσου σημαντικό να πετύχουμε μεγαλύτερη συνολική συμμετοχή, καλύτερη υλοποίηση και ε, συμμόρφωση με αποφάσεις και υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Και εδώ βρίσκεται και η σημασία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας. Διότι με μια καλύτερη δομή οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της λέσχης των 20 μπορούν να βρουν την νομιμοποίησή τους με τη διαφάνεια και την υλοποίηση μέτρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπογραμμίζουμε στην έκθεση την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ομιλεί με μια ενιαία ισχυρή φωνή. Την ανάγκη να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενδυνάμωση, στην ενίσχυση της ε, οικονομικής διακυβέρνησης ε, και του παγκόσμιου πρωτοπόρου ρόλου που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο, τον κύριο Χέκμαρκ, για την ε, έκθεσή του και τα σχόλιά του. Δύο πράγματα θέλω να πω μόνο. Πρώτον, ε, ο φόρο επιχρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που, στον οποίο αναφέρθηκε όλο ιδιαίτερο ο πρόεδρο Μπαρό ω κάτι ευκταίο και ω κάτι πρέπει να εφαρμόσουμε στην Ευρώπη ή τουλάχιστον στην Ευρωζώνη, νομίζω ότι είναι προφανώς ένα λεπτό θέμα Νομίζω ότι είναι λογικό, είναι δίκαιο. Ο χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να συνεισφέρει, γιατί έχει πάρει ήδη 3,5 δισεκατομμύρια από χρήματα των φορολογουμένων, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί αλλιώ ε, θα ε, οδηγηθούμε σε στρέβλωση των επενδύσεων σε διάφορα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεύτερον, συμφωνώ απολύτω με τον κύριο Μάρκο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία φωνή θα πρέπει να μιλάει και αξίζει την ιδιότητα του μέλους ε, του ΠΟΕ, την ψήφο της ε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σίγουρα που να επικρατήσει διαφάνεια σχετικά με την εκλογή του εκτελεστικού διευθυντή. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπαζέσκου. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χεκμακ πρώτα απ' όλα για αυτή την έκθεση. Η έκθεση καταδεικνύει την ανάγκη της παγίωσης ε, και εδραίωσης ε, της ε, παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Η απουσία συντονισμού σε αυτά τα οικονομικά συστήματα θα μπορούσε να συνεπάγεται απουσία λύσεων στα προβλήματα. Το σύστημα όμως πρέπει να βελτιωθεί με την εισαγωγή νέων ελεγκτικών μηχανισμών και ρυθμίσεων και διατάξεων. Δυστυχώς ε, βλέπουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η συνάντηση της Λέσχης των 20 είναι απλώς και μόνο μέσα τα οποία όργανα τα οποία έχουν περιορισμένες ε, εξουσίες και αρμοδιότητες. Χρειαζόμαστε όμως μια σφαιρική ολοκληρωμένη λύση για αυτά τα προβλήματα και την κρίση. Η χώρα μου έχει εισαγάγει και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε ο απολογισμός ο αρνητικός να μειωθεί και το έλλειμμα να μειωθεί μέχρι το 2012. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα. Όταν κάνουμε λόγο όμως για τις ε, παγκοσμιοποιημένες, παγκόσμιες πτυχές για την οικονομική διακυβέρνηση και τα αποτελέσματα της λέσχης ε, των 20, της συνάντησης της λέσχης των 20, αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα χειροπιαστά, πρέπει να προβληματιστούμε για την ευρωπαϊκή συνιστόσα. Δυστυχώς φαίνεται ότι με πολύ βραδείς ρυθμούς ε, καταλήγουμε στην ε, υιοθέτηση λύσεων ε, στην Ευρώπη. Αυτό αφορά και την ελληνική κρίση και αυτό οδηγεί στο να εγκυμονούν πάρα πολύ κίνδυνοι και για την Ευρώπη και παγκόσμια. Δεν υπαρκούν όλα αυτά. Γι' αυτό είναι χαρμόσυνο το ότι αυτή η έκθεση πηγαίνει πιο πέρα από τα ισκαμένα και δίνει κίνητρα για να σημειωθεί πρόοδος. Επειδή έχουμε ακριβώς την επιτυχή οικονομική πολιτική και άλλες λύσεις που προτείνονται στην οικονομική διακυβέρνηση σε παγκόσμιο πλαίσιο. Η σταθερότητα όμως του Ευρωπαίου να διασφαλιστεί. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, τότε δεν θα έχουμε και αποτελέσματα ακόμα και στις συνόδους κορυφής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ο κύριος Χεκμάκ συνέταξε την έκθεσή του και είναι πολύ καλή η έκθεσή του πριν από τη Σύνοδο Κορυφή τη Λέσχη τον 20 τον Νοέμβριο, πολλά πρέπει να πράξουμε στο επίπεδο, στον τομέα τη ε, παγκοσμιοποιημένη οικονομική διακυβέρνηση. Δύο πράγματα ε, εν συντομία θέλω να αναφέρω. Οι εμπλεκόμενοι, οι περισσότεροι από εμπλεκόμενου γνωρίζουν το υφιστάμενο οικονομικό σύστημα ότι αποσυναρμολογείται, αποξυλώνεται και δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Κατανοούμε λοιπόν αυτή την έκθεση ως μια καλή έκθεση επειδή η κατάσταση είναι απαράδεκτη ως έχει. Όμως ακόμα είναι ασαφές αν ένα νέο σύστημα το οποίο θα αναδυθεί από τα ερήπια του παλαιού αν ένα τέτοιο νέο σύστημα θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Γιατί αν υπάρξουν αρνητικές ε, εξελίξεις ε, σαν συνέπεια αυτής της αναδόμησης η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ζητούμε οι Ευρωπαίοι και οι παγκόσμιοι οι ηγέτες να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να δράσουν αντίστοιχα, διότι πρόκειται εδώ για τους ίδιους τους πολίτες και την επιβίωση. Σικλούνα, ο κύριος Σικλούνα. Πρόεδρε, ε, η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζουν ένα βέβαιο μέλλον ε, και άρα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό το θέμα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της Συνόδου για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας ε, των 20. Ε, στην έκθεση του κυρίου Χιωεκμάρε τονίζονται οι ανισορροπίες και νομίζω θα πρέπει οι θυνοντές να λάβουν υπόψη αυτά τα μηνύματα. Τι χρειαζόμαστε, συνεργασία ανάμεσα στις χώρες, ούτως ώστε να επιτύχουμε την οικονομική ανάκαμψη και να συναυτούν εμπορικές συμφωνίες. Και η G20 και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι οι δύο βασικότεροι φορείς στην παγκόσμια οικονομία, θα πρέπει να εξασφαλίσουν μηχανισμούς σταθερότερης οικονομικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ώστε να ακούγεται και η φωνή των BRICS, ε, το οποίο θα απηχεί και την οικονομική πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε επίση μια κρατεία νομική βάση, ώστε να είναι ε, ε, δεσμευτικέ οι αποφάσει του. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των διεθνών οικονομικών φορέων. Χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα, ούτω ώστε να γίνονται επενδύσει σε Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι αλληλένδετες σε όλες τις οικονομίες και θα καταρρύψει ολόκληρο το σύστημα αν δεν κάνουμε κάτι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερέιρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το βασικό θέμα ε, που αποφεύγει και η έκθεση και η συζήτηση είναι οι αιτίε ε, αυτών των παγκόσμιων ανισορροπιών. Ποιε είναι οι πραγματικέ αιτίε ε, τη παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν φέρουμε στη συζήτηση. Από ό,τι φαίνεται επιμένουν κάποιοι να συνεχίσουν στον δρόμο που μας οδήγησε μέχρι εδώ ε, και μας παρουσιάζουν την ανάγκη ως επιτεκτική για να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία της ε, οικονομικής καταστροφής. Φυσικά ζούμε μια κρίση, την κρίση του καπιταλισμού, όπου ε, την κρίση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και η λύση δεν θα προέλθει από τους ε, διεθνικούς οργανισμούς ε, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις τους να συνεχίσει η παραγωγή στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος ε, παραβιάζει την κυριαρχία και τη δημοκρατία των κρατών μελών παραβιάζοντας τα δικαιώματα όλων η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων η απελευθέρωση του παγκοσμίου εμπορίου είναι η, η μια ταινία που έχουμε ήδη δει όλοι γνωρίζουμε πώς τελειώνει αυτή η ταινία. Ε, γνωρίζουμε ανισορροπίες και αδικίες σε ε, παγκόσμιο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί αν αφήσουμε τις αποφάσεις σε αυτούς τους ε, διεθνείς οργανισμούς που έχουν καταδείξει ότι σίγουρα δεν είναι καλοί φίλοι και δεν πρέπει καν να τους αναστρεφόμαστε. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Χέκμακ στην αναφορά του ότι είναι αναγκαίο, όπως είπε, να συζητήσουμε για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και το σύστημα που θα ακολουθηθεί στη συνάντηση της Λέσχης των 20 διότι ακριβώς εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον και τον συντονισμό για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την οικονομική διακυβέρνηση. Και δεν, είμαι, δεν έχω τη βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή μπορεί να προσφέρει πραγματικές εναλλακτικέ λύσεις, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να τα επιλύσει η ίδια. Και μπορούμε να θυμηθούμε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 πρόσφατη οικονομική κρίση και τα αίτια της ρίζες αυτής της κρίσης ε, που εξακολουθούν να μην έχουν αντιμετωπιστεί και να μην έχουν επιληθεί και θα πρέπει οι ηγέτες μας να βρουν επικοδομητικές λύσεις στα προβλήματα που κλειδονίζουν και κλονίζουν τη σημερινή Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αναμένουμε λοιπόν η, ο, ο, η παγκοσμιοποιημένη κοινότητα να αφουγκραστεί, να τίνει ευήκονους στους Ευρωπαίους πολιτικούς που δεν έχουν μπορέσει να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος έχει το λόγο, κύριε Ρέντινγκ. Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να καταθέσουν αυτή την εβδομάδα ε, δυνατές προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να εξέλθουμε από την κρίση του. Του λεκθέντος σωστά τονίζει ο κύριος Χέκμαρ την σημασία της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης που συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση των εθνικών προβλημάτων σε όλες τις υπήρους. Και ενστερνιζόμαστε πολλές από τις συστάσεις του κύριου Χιόκμερ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους βουλευτές που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τους ευχαριστώ για τη συνεισφορά τους. Η τωρινή κρίση οδήγησε σε βαθιά κρίση και της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Πριν το 2008 δεν είχε ε, σκεφτεί κανείς ότι θα σημειωνόταν μεγάλη πρόοδος για την σύγκληση των οικονομιών ή ότι επρόκειτο να δώσει απάντηση η ομάδα των 20 πλουσιότερων χωρών για την ε, ύφεση και την ε, επιβράδυνση οικονομικής δραστηριότητας. Συνέβησαν όμως όλα αυτά και τώρα έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ διεθνούς οικονομικής συνεργασίας αυτή η λέσχη. Όμως δεν φτάνει αυτό. Χρειαζόμαστε ε, και άλλα μέτρα για να για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιβράδυνση, της, ε, την ύφεση της οικονομίας ε, χρειά και εντός ολίγου σας είπα ότι θα καταθέσουμε προτέσεις. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να προσθέσω θα έπρεπε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα για να το κάνουμε αυτό και αυτό έχουν κατά νου αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και αυτό θα πράξουν. Ε, την τρέχουσα εβδομάδα ο Πρόεδρος Μπαρόζο στην ε, ομιλία που έκανε ενώπιον του Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ένωσης είπε ότι ήρθε η στιγμή να έχουμε μία ενοποιημένη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετόνωση της εσωτερικής οικονομικής διακυβέρνησης και μου έρχεται κατά νου η δέσμη των έξι οδηγιών Τώρα θα πρέπει να οδηγηθούμε και προς μια ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση κατά πρώτο λόγο στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σύντομα θα καταθέσουμε προτάσεις για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Τελειώσαμε με αυτή τη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Τώρα, έκθεση ματέρα για την κατάσταση των